Το πρώτο θέμα. Έκθεση Ματίας. Έρευνα και καινοτομία και σχετική χρηματοδότηση. Αυτή είναι η πρώτη συζήτηση. I not all of you καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε όλοι να μείνετε στην αίθουσα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εγκαταλείψετε συντόμως στην αίθουσα και να μην συζητάτε εντός αυτής. Έχετε διαδικαστικό. Διαδικαστικό. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως θα ακολουθήσω την ε, πρότασή σας. Θα μείνω εγώ στην αίθουσα, αλλά σας παρακαλώ να μην βλέπετε μόνο ευθεία μπροστά, αλλά να δείτε δεξιά και αριστερά. Γιατί είναι ε, πάρα πολύ δύσκολο να ζητάει κανείς τον λόγο και να μην μπορεί να πιάσει το μάτι σας γιατί δεν μπορείτε να κοιτάτε προς όλες τις κατευθύνσεις. Παρακαλώ λοιπόν να ρίχνετε μια ματιά και σε μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το έχω κατά νου, κυρίες και κύριοι. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Ματίας, η οποία είναι η συγκήτρια για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της έκθεσης και κυρίως να σας ευχαριστήσω γιατί ήταν μια περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη. Ήταν η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών. Παρ' όλα αυτά όλοι ήταν διαθέσιμοι για να συνεργαστούν στην επεξεργασία συμβαστικών λύσεων και έτσι σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε ε, με όλους ε, το περιεχόμενο της ε, έκθεσης. Ευχαριστώ για τις γνωμοδοτήσεις επίσης από τις διάφορες επιτροπές που συνέβαλαν, γνωμοδοτήσεις που εντάχθηκαν στην τελική έκθεση. Και πριν να περάσω στο ίδιο το περιεχόμενο της έκθεσης δεν μπορώ παρά να ε, εκφράσω την εκτίμησή μου και τους, τους δύο υπαλλήλους, Σουζάννα Κίφερ και Γιώραν Γκάιν των Επιτροπών ε, Βιομηχανίας που, της Επιτροπής Βιομηχανίας που έμειναν να δουλέψουν και τις καλοκαιρινές διακοπές. Πρόκειται για μια στρατηγική για την καινοτομία και την τεχνολογία για την περίοδο 2014 με 2014. Είχαμε ευκαιρίες να το συζητήσουμε το θέμα επανελειμμένως και με την ε, Επίτροπο. Κατά τη γνώμη μου είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να τονίσουμε την προστιθέμενη αξία των, ε, της δικής μας τεχνολογίας και τενοτομίας. Το κοινό πλαίσιο χρηματοδότησης για την καινοτομία και την ε, τεχνολογία δεν μπορεί να γίνει μόνο με μεμονωμένες προσπάθειες. Γι' αυτό και στο πρόγραμμα πλαίσιο το να συνδεθεί με αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, να συνδεθεί επίσης το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, καθώς και όλα τα ποσά ε, τα οποία έχουν χορηγηθεί για όλα αυτά τα προγράμματα. Δεν έχουμε μια κοινή στρατηγική, δεν θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε ε, και να επιτύχουμε τους στόχους. Και γι' αυτό εξ αρχής θα ήθελα να μιλήσω για τους βασικούς στόχου στόχους. Πιστεύω πως τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας βασικά εξυπηρετούν τρεις βασικές διαστάσεις. Καταρχήν την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ερευνητών της Ευρώπης που είναι ο πιο σπουδαίος πόρος που έχουμε για την έρευνα. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους μέσω της ενίσχυσης των υποδομών είναι απαραίτητη επένδυση που πρέπει άμεσα και κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε το δυναμικό συνεργασίας που έχουμε στον τομέα της ε, έρευνας. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί αυτός ο τομέας ώστε η καθοριστική τομή για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας όπως οι κοινωνικές επιστήμες χωρίς αυτές δεν μπορούμε να έχουμε καινοτομία, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την κοινωνία στην οποία θα πρέπει να παρέμβουμε από πολιτικής άποψη και γι' αυτό δεν μπορούμε και να τι εγκαταλείψουμε. Και έπειτα έχουμε και την καινοτομία και την, ε, τον προσανατολισμό αυτής προς την αγορά. Το να ορίσουμε κοινού στόχους μέσα στο κοινό πλαίσιο θα εξυπηρετήσει όλους και θα εξυπηρετήσει και την έρευνα και την τεχνολογία ώστε να γίνουν καθοριστικοί παράγοντες σε μια περίοδο τόσο σημαντική όπως αυτή που διανύουμε τώρα, την οικονομική και κοινωνική κρίση, τη χρηματοπιστωτική κρίση όπου διαρκώς μεγαλώνουν οι αποκλήσεις και τα κενά. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει συνδυασμό μεταξύ των διορθωτικών ταμείων και είναι πολύ σημαντικό να απλοποιηθούν τα διάφορα μέτρα ώστε να μπορέσουν οι ερευνητές να ε, χρησιμοποιήσουν τα γραφειοκρατικά ε, συστήματα που υπάρχουν στη διάθεσή τους σε μια Ευρώπη αποκλήσεων, ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να αποτελεί έναν αγώνα όπου πάντοτε θα κερδίζουν μόνο αυτοί που έχουν ε, πρόσβαση στα κονδύλια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εγγυηθούμε, κυρία Επίτροπε, και το γνωρίζετε κι εσείς, ο ανταγωνισμός να είναι θεμητό, υγιής, μέσα στις καλύτερε δυνατές συνθήκε, αλλά μέσα στο πλαίσιο σύγκλησης στην Ευρώπη να γίνει μια περιοχή αριστεία. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Θα ήθελα να ζητήσω εξ ονόματος της Επιτροπής να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Μέγερ Γκόγεν Κουίν. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω πριν από την τελική ψηφοφορία αύριο επί της ε, Πράσινης Βίβλου για το κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ένωση, που τώρα είναι γνωστή ως πρόγραμμα 2020. Συγχαίρω την κυρία Ματίας για το ότι έγραψε μια πάρα πολύ έκθεση και εγκαίρος και επέτρεψε έτσι η Κομισιόν να δει την πρότασή της εις ε, βάθος στο πλαίσιο του πακέτου 2020. Επίσης να ευχαριστήσω τους και ηγητέ της Επιτροπής Ήτρε και των έξι επιτροπών που έδωσαν γνωμοδοτήσει στο Κοινοβούλιο επέδειξε τρομερό ενδιαφέρον για τη λειτουργία του μελλοντικού πλαισίου στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς θα σας αποστείλουμε σύντομα τις προτάσεις για τον ορίζοντα του 2020, που βεβαίως οι προτάσεις αυτές ελοποιηθούν από το νέο χρηματοοικονομικό ορίζοντα του 2014. Έχουμε έτσι το πολιετές πλαίσιο το οποίο ευθύθηκε 29 Ιουνίου και έχουμε συνολικό προβλησμό 80 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τιμές 2011. Ο προπολογισμό αυτός έχει στόχο να προωθεί στην ανάπτυξη και τις ε, δουλειές. Ο συνολικός αυτός φάκελος είναι ρεαλιστικός και φιλόδοξος και το να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτές τις επενδύσεις τώρα θα μας επιτρέψει να έχουμε ανάπτυξη και δουλειέ στο μέλλον. Με αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει σαφώς την δέσμευσή της για να έχει αποτελέσματα στις φιλοδοξίες της Ευρώπης 2020 και μια ένωση της καινοτομίας. Ο στόχος του ορίζοντα 2020 είναι να γίνει πιο αποτελεσματική η χρηματοδότηση της έρευνας με πιο εύκολη πρόσβαση και να έχει περισσότερα αποτελέσματα. Η συντριπτική απάντηση στην διαβούλευση ήταν ναι, μια πάρα πολύ πρακτική συνεισφορά στο πώς θα το επιτύχουμε αυτό. Είχαμε πάνω από 1.300 απαντήσεις και υπευλήθησαν επίσης 750 προτάσεις. Θα ήθελα τώρα να να ευχαριστήσω την κυρία Ματίας και όλους τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην εκδήλωση της 10ης Ιουνίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης. Ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για να δείξουμε στους ενδιαφερομένους πως τα θεσμικά όργανα της Ένωσης συνεργάζονται για να επιτύχουν τους ίδιους στόχους. Νομίζω πως τα βασικά ζητήματα είναι τα ίδια με αυτά τα οποία ετέθησαν στην διαβούλευση. Συμφωνούμε σε γενικές γραμμές για τα βασικά ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε θα ήθελα να τονίσω κάποιες από τις προτάσεις για τον ορίζοντα 2020 που είναι πολύ ενδιαφέρουσες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με την ισχυρή στήριξη που δείχνεται για την έννοια του κοινού στρατηγικού πλαισίου και το πώς θα έρθει πιο κοντά η στρατηγική της έρευνας ε, και της καινοτομίας και πώς θα πάμε από το εργαστήριο στην αγορά. Η αριστεία θα παραμένει το βασικό κριτήριο κατανομής των χρημάτων, ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες οδούς προς την αριστεία για τις περιοχές και τις χώρες εκείνες οι οποίες υποεκπροσωπούνται. Και αυτό βέβαια είναι αρμοδιότητα των διαρθρωτικών ταμείων. Θα πρέπει οι ερευνητέ μα να εργάζονται περισσότερο και να μην ασχολούνται με τα διοικητικά. Η απλοποίηση θα είναι βασικό στοιχείο του πακέτου ορίζοντα 2021 σημείο στο οποίο συμφωνούμε είναι πως θα πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια όσον αφορά τα επιτυχή μέσα του προγράμματος. Και εδώ πέρα μιλάμε κυρίως για την συνεργασία στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο Έρευνα και τις δράσεις Marie Curie. Χαίρομαι για το ότι υποστηρίζουμε το ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση της Ένωσης να είναι κοντά στι προκλήσει κοινωνία, όπω παραδείγματο χάρη κλιματική αλλαγή, υγεία και ενεργειακή ασφάλεια. Θα ήθελα επίση να τονίσω πω η έκθεση Ματία συμπεριλαμβάνει πάρα πολλέ ιδέε που προβλέπονται ήδη στην έκθεση Καρβάλιο περί απλοποίηση, την έκθεση Μαρκή για την Ένωση Καινοτομία και την εκθέση ΟΝΤΗ για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 από την σκοπιά τη Κομισιόν. Η συνέχεια και η συνέπεια έχει διατηρηθεί και αυτό μα βοηθάει πάρα πολύ καθώ προετοιμάζουμε τι νομοθετικέ προτάσει για τον ορίζοντα του 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κουίν, κυρία Επίτροπε και συμπαθάτε με διότι δεν πρόφερα σωστά το όνομά σα, το επώνυμό σας. Κολίκ. Καρλ uh, από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ. Θεωρώ πως το τελικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Ε, τα όσα θα ψηφίσουμε αύριο, κυρίως όσον αφορά το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το οποίο μίλησε και η Επίτροπος. Κάτι ακόμα που πρέπει να τονίσουμε όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές ε, επενδύσεων είναι ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τον οποίο εμείς βλέπουμε ως πολύ θετικό. Επιπλέον υπάρχει και το θέμα της διαφοράς ανάμεσα στις ε, υποτροφίες και τις ε, αμοιβέ. Όσον αφορά την ε, στρατηγική 2020 γνωρίζουμε πως θα είναι δύσκολο να καταφέρουμε να συλλέξουμε τους πόρους και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κινητοποιηθούν και τα ταμεία, το Ταμείο Συνοχής. Επιπλέον θα πρέπει να αποφευθύνουν τα προβλήματα όπως ε, η χρηματοδότηση του ΙΤΕΡΑ για να μην ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λάρα Κόμη από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και, Κατανάλωση, και Καταναλωτή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε αυτήν την έκθεση εντοπίζουμε πολλές σημαντικές πτυχές που θα πρέπει να ληφθούν ε, καταλήλως υπόψη. Ο συντονισμός ανάμεσα στα προγράμματα καινοτομίας και τεχνολογίας, τα ταμεία συνοχής μέσω της ενίσχυσης του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών αρχών, επιπλέον απλοποίηση της διαδικασίας και ευελιξία που είναι απαραίτητη για την ενημέρωση των προγραμματικών προτεραιοτήτων η χορήγηση ενός κομματιού των κονδυλίων για τους νέους και τις νέες ε, ε, επιχειρηματίες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω κάτι που εγώ προσωπικά τόνισα και που σημαίνει ε, ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί μέσα στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο ένας πειραματισμός που θα βασίζεται στην αρχή της πιστοποίησης ώστε οι επιχειρήσεις να προσανατολιστούν στην τεχνολογία τεχνολογική και καινοτόμα ανάπτυξη έτσι ώστε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια να μπορούν δραστήρια να συμμετέχουν σε καινοτόμες ε, διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Έρμαν Ίνκλερ, από όσο ξέρω δεν είναι εδώ, ο, κύριο, ο κύριος Τζοβάνι Λαβία. Σας ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, και στην ε, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπέθρου θελήσαμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει η έρευνα για ολόκληρη την προοπτική του, αγρο, τον, ε, τομέα των ε, γεωργικών, γεωργικής παραγωγής και τροφίμων. Μπορεί να μετατράψει συγκεκριμένα σε έρευνες σε αποτελέσματα επιτόπου. Μπορέσαμε να υπογραμμίσουμε πως η έρευνα θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στους πολίτες του κόσμου. Έχουμε μια αυξητική προοπτική στον πληθυσμό, έντονη προοπτική, το 70% επιπλέον θα ζητά ε, τρόφιμα μέχρι το 2050. Και θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά όλα και μέσω της έρευνας που θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξει όλο ένα και περισσότερο και τις ανάγκες για ένα καθαρό περιβάλλον. Πρέπει να συνδυάσουμε δηλαδή την αύξηση της παραγωγής με την προστασία του περιβάλλοντος, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιωάννης Τσουκαλάς, Επιτροπή Ελίας. President, αναπληρωματικό μέλος της ΠΕΣ, εκπροσωπώ τον συνάδελφο κύριο Βαλένσα, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί στην παρούσα ολομέλεια. Η παρούσα έκθεση είναι εξαιρετική σημασίας για την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και καινοτομίας καθώς επιχειρεί να περιορίσει επικαλύψεις και σπατάλες και να θέσει ενιαίους ευρωπαϊκούς στόχους και μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένες δυστυχώς και της δικής μου εξακολουθούν να απέχουν πολύ από την επίτευξη του στόχου του 3% του ΕΠ για την έρευνα και την καινοτομία έως το 2020, γεγονός που αναμφίβολα οδηγεί σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Και όταν φυσικά μιλούμε για το έλλειμμα στην έρευνα, δεν ανοούμε μόνο τους τομείς της υψηλής τεχνολογίας. Ιδιαίτερα σημαντική, αν και όχι προφανής, είναι η ανάγκη για στήριξη της έρευνας στον τομέα της αλίας δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον παραμελημένο τομέα της αλληλείας μπορούν να διαμορφώσουν ένα πιο ανταγωνιστικό βιώσιμο σύγχρονο αλλιευτικό κλάδο και να ωφελούσουν σημαντικά τους Ευρωπαίους που εξαρτώνται από την αλλιευτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, dziękuję ε, Ponieważ wspomniał pan pana Jarosława Wałęsy, naszego kolegi, który nie mógł wystąpić dzisiaj przed Μιλήσατε για τον ε, συνάδελφο Βαουέζα που δεν είναι παρόν στην αίθουσα. Τον επισκέφθηκα στο νοσοκομείο. Ήθελα να σας πω ότι περασμένο Σάββατο ε, μου είπε πως ε, το αργότερο το Μάρτιο θα είναι κοντά μας και ίσως και το Φεβρουάριο υγιής και σας διαβάζει τους χαιρετισμού του και τις ευχές του σε όλους τους συναδέλφους του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας διαβιβάσω το την ευχή του. E, Το λόγο έχει τώρα η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου από την Επιτροπή Γυναικών. Ω Επιτροπή Γυναικών, θεωρούμε πω η γυναικεία επιχειρηματικότητα εξασφαλίζει δυναμισμό και καινοτομία στι επιχειρήσει και συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού απασχόληση των γυναικών, που είναι από του βασικού στόχου τη στρατηγική Ευρώπη 2020 ωστόσο υπάρχουν αναξιοποιητέ γυναικείε εφεδρείε στον τομέα τη έρευνα και τη καινοτομία οι γυναίκε ερευνήτριε βιώνουν δυσμενεί διακρίσει πάγια στερεότυπα τα φαινόμενα τη γυάλινη οροφή και τη διαρροή αγωγού ανεπαρκή χρηματοδότηση και άνισε ευκαιρίε ανέλυξη. ζητούμε λοιπόν την ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο και σωστή χρησιμοποίηση διαρθρωτικών ταμείων και πολιτικών συνοχή ώστε οι γυναίκε ερευνήτριε να αναπτύξουν καινοτόμα επιχειρησιακά προγράμματα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιστημονικά επιστημονικά προγράμματα να έχουν επαρκή κινητικότητα και να συμμετέχουν σε πλατφόρμες δικτύωσης. προτείνουμε τέλος να προβλεφθεί ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων ως μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που να διασφαλίζει ακριβοδίκαιη κατανομή χρηματοδοτήσεων στη βάση έρευνας δικτών και στοιχείων του ευρωπαϊκού συμβουλίου έρευνας. ευχαριστώ. Τώρα ακολουθούν οι μιλητές ε, εξ των κομμάτων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, κυρία Καρβάγη. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την ε, βουλευτή Μαρίζα Ματίας για την εξαιρετική της εργασία και για την οικοδομητική της συνεργασία με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ε, η ομάδα του ΕΛΚ είδε πως οι βασικές του προτάσεις συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση, αύξηση δηλαδή του, επομένου, του προπολογισμού του επόμενου πλαισίου για την ε, καινοτομία και την τεχνολογία, συντονισμός με το πόρους από των διευθυντικών ταμείων, η συμπεριλήψη του δρόμου για την αριστεία, η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την καλύτερη εξέλιξη των, των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, συμμετοχή των νέων ερευνητών, απλοποίηση τον... Ε, διαδικασιών. Είναι δύο πυλώνες για την ανάπτυξη, την οικονομική και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι γι' αυτό σημαντικό να αυξηθεί το τμήμα της χρηματοδότησης που δίνεται στην έρευνα και στην τεχνολογία μέσα στην πλαίσιο της σημαντικής αύξησης του προγράμματος πλαισίου και του ποσοστού των διευθυντικών ταμείων που αφοσιώνονται, αφιερώνονται σε αυτό το τομέα. Ο πρώτος στόχος του προγράμματος πλαισίου είναι να προωθήσει την αριστεία και θα να εξακολουθήσει να είναι αυτό ο πρώτο στόχο, αλλά είναι επίση σημαντικό να δημιουργηθούν απαραίτητε προποθέσει για τη συμμετοχή μικρών μονάδων, κέντρων αριστεία, με, με, με μικρέ ερευνητικέ ομάδε και καινοτόμε επιχειρήσει. Έχοντα αυτόν τον στόχο, η έκθεση προτείνει Δούσου για την αριστεία γνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο του επιχειρηματικού ιστού στην ανάπτυξη, την οικονομική και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, το ΕΛΚΑ είναι ευχαριστημένο με το ότι όλα αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση. Οι νέοι επίσης με ψηλές, ψηλά προσόντα να μπορούν να κινηθούν στην Ευρώπη, κάτι που θα είναι προς όφελός τους. Τέλος, η απλοποιημένη πρόσβαση στους πόρους για την έρευνα για να δημιουργηθεί μια νοοτροπία εμπιστοσύνη σε όλους τους συμμετέχοντες ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η τεχνολογία στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Έρτσογκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή εργασία. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέτουμε μεγάλους στρατηγικούς στόχους και να τους διατυπώνουμε. Πρώτος αυτός στόχος θα μπορούσε να είναι για εμάς σοσιαλιστές να έχουμε αυτό το πολιετές πρόγραμμα των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ να το δούμε ως μια επένδυση και όχι ως χρήματα τα οποία θα υποκαταστήσουν άλλες πηγές ε, χρηματοδότησης. Και πρέπει να πολλαπλασιαστεί, μάλιστα, να μην πω τετραπλασιαστεί αυτό το ποσό. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του 2020 υπάρχουν και άλλες υποπροτεραιότητες, όπως παραδείγματο χάρη η έρευνα, την οποία θα πρέπει να έχουμε κατά νου αν θέλουμε έξυπνες τεχνολογίες, πράσινες τεχνολογίες, ε, θα πρέπει να κάνουμε και ανάλογα βήματα. Το τρίτο στόχος είναι η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι ερευνητές μας ε, να μην χρειάζεται να μετακομίζουν βόρεια και δυτικά αλλά να μπορούν να παραμένουν στα δικά τους κράτη-μέλη για να εκμεταλλευτούν το ταλέντο τους. Επιπλέον χρειαζόμαστε μια νέα βιομηχανική πολιτική. Ξέρετε, τα αποτελέσματα εκείνα της καινοτομίας ε, τα οποία υπάρχουν θα πρέπει να δημιουργούν περισσότερα πράγματα σε μια κάθετη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως η κυρία Εκ δεν είναι εντός αιθούσης, οπότε δίνω το λόγο για ένα λεπτό στην κυρία Σουίνμπορν. Θα πρέπει η χρηματοδότηση αυτή να ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο που να βοηθούμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, γιατί πάρα πολύ συχνά οι εταιρείε αναφέρονται στις αντιφατικές μας πολιτικές και την να εβδομάδα γίνεται το ίδιο όσον αφορά τα ταυλά στο κύτταρα και τη χρηματοδότηση. Ε, γιατί οι έρευνε θα πρέπει να είναι αναλλακτική λύση στι δοκιμέ ζώα. Αυτό όμω θα πρέπει να το αγκαλιάσουν όλα τα κράτη-μέλη και ε, λένε όλες οι εταιρείε ε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μη αντιφατικές πολιτικές, οπότε θα είναι δυνατόν να έχουμε τελικά κάποιο είδους αποθετήριο, θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των βασικών ε, παραγόντων και των ακαδημαϊκών αρχών για να έχουμε επομένω παγκόσμιες κλάσεις έρευνα για να μείνουμε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να μπορούμε συνεχώς να έχουμε κάποιο είδου ε, αυτοέλεγχο από τους εμπλεκομένους. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Τώρα, ο κύριος Λαμπέρτς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την κύριε Επίτροπο και εμείς όπως και εσείς ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλη επιτυχία αυτό το οποίο καταφέρατε, ολοκληρώσαμε τον προβληματισμό για τα δημοσιονομικά σε σχέση με αυτό το θέμα το οποίο είναι σημαντικά βελτιωμένο γιατί έχουμε δύο βασικές ε, επιτυχίες όσον αφορά ε, το να έχουμε αποτελεσματική έρευνα για καινοτομία στην Ευρώπη. Ε, Θα να σας πω ότι να προσέξουμε την απλούστευση, διότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η διοίκηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει απλουστευμένες διαδικασίες. Αλλά αυτό κυρίως αφορά τους τελικούς χρήστες και τις επιχειρήσεις αυτοί οι οποίοι απευθύνονται στις θηρίδες της Επιτροπής, διότι κυρίως για αυτούς θα πρέπει να έχουμε μια προστατευμένη διαδικασία. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε όμως στο στον ούτω υπήν πελάτη και όχι να έχουμε εσωστρέφει στις διαδικασίες μας, κάτι, κάτι άλλο τώρα, να μπορέσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας να τα μεταλαμβαδεύσουμε στην ε, αγορά και να είμαστε και στην κοινοτομία όπως και στην ερευνά το ίδιο καλή. Εδώ επιδέχεται η βελτίωση η κατάσταση και επίσης δεν θα πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο ε, να προσέξουμε μόνο την καινοτομία. Και έτσι με συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα ή μέσω αμέσων επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις να δούμε πώς δεν ε, θα δικήσουμε ε, η κατάσταση βοηθώντας εταιρείε που έτσι και αλλιώς μπορούν και έχουν τα μέσα να κάνουν επενδύσεις. Άρα ε, να μην βοηθήσουμε αυτούς που δεν έχουν ανάγκη τη βοήθεια για την καινοτομία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ένιν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ένωση βλέπει την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας που έπρεπε να καταστήσει την Ευρώπη την οικονομία γνώσης την πιο ανταγωνιστική και την πιο δυναμική του κόσμου για το 2010. Η Κίνα και όχι η Ευρώπη θέτει σε εφαρμογή του στόχου της στρατηγικής της Λισαβόνας. Το 2010 οι δαπάνες ιδιωτικές και οι δημόσιες της Κίνας έφτασαν αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σύντομα η Κίνα θα έχει περισσότερους μηχανικούς και ερευνητές από ότι η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από σε αυτό το πολύ εντυχητικό πλαίσιο μόνο ο τομέας της ε, ευρωπαϊκής Αεροπλοεία υπάρχει και επιζεί ακόμα γιατί η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία μπόρεσαν να αναλάβουν τις ευθύνες του επενδύοντα ε, στο μακροπρόθεσμα και σεβόμενοι το δόγμα ε, της ελεύθερου ανταγωνισμού. Ε, τα ισχνά επιτεύγματα της ευρωπαϊκής έρευνας ε, είναι, οφείλονται στην λάθος βιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Είμαστε ακόμα κάτω και από τη διάγνωση των αιτίων και των λύσεων για αυτή την κατάσταση, την ανησυχητική. Αυτό που είναι στην καρδιά του προβλήματος είναι η έλλειψη δημοσίων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας Επίση, ε, είναι γεγονό ότι οι νέοι ερευνητέ και οι μηχανικοί είναι πολύ επισφαλεί στι θέσει του και κακοπληρωμένοι. Ενώ οι traders ε, τη οικονομία ε, αμείβονται σκανδαλωδώ πολύ. Είναι πρίμα εγκλήματα αυτά. Η έλλειψη των επενδύσεων στην ανάπτυξη μια επιστημονική και τεχνική μαζική νοοτροπία από την πιο μικρή ηλικία είναι το αίτιο. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί η γνώση και η τεχνογνωσία στην Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μα έδειξε ποιο είναι το όραμα όσον αφορά το καινούργιο στρατηγικό πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογία, σχετική χρηματοδότηση για την περίοδο που θα ακολουθήσει το 2013, διότι κάθε επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στις ε, χώρες ε, της Ένωσης ε, πάει τώρα στο 1,5 του ΑΕΠ. Άρα είμαστε πολύ πίσω από τους ανταγωνιστέ μας και μέχρι σήμερα η πολιτική που ακολουθούμε δεν μας έχει οδηγήσει σε κάποιες βελτιώσεις. Άρα θα πρέπει να θεωρήσουμε το σύστημα και θα πρέπει να βοηθήσουμε έρευνα και καινοτομία. Υπάρχουν μια σειρά προτάσεων εδώ, όπως και αυτή την, την, την ε, προσέγγιση των τριών βημάτων, όπως είπε η κυρία Μαρίσα Ματίας, η συγκήτρια, ούτως ώστε να άρουμε τους φραγμούς που εμποδίζουν τις ε, ΜΜΕ να έχουν προσβασιμότητα στη χρηματοδότηση. Θέλουμε κάποιε διαδικασίε ενταγμένε σε όλε τι πολιτικέ, ούτω ώστε ο κόσμο να αποφαρύνεται από την γραφειοκρατία. Και οι εφευρέσει όμω θα πρέπει να γίνονται προϊόντα όσο γίνεται συντομότερα. Και έτσι να βοηθήσουμε την έρευνα στην Ευρώπη που θα πρέπει να αποδώσει αποτελέσματα όσο γίνεται πιο γρήγορα διότι όπως είπαμε ε, έχουμε μείνει πίσω και αυτό είναι παράδειγμα. Ευχαριστώ για πρόεδρος. Ρόιλ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω την ε, κυρία Ματίας ε, και τους συναδέλφους που προηγήθηκαν, κυρία Μερικής και Καρβάλιο και υπάρχει εδώ πέρα μία συνέχεια. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει όχι μόνο να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις, αλλά να αποδείξουμε ότι παίρνουμε σοβαρά τα ζητήματα της έρευνα και της καινοτομία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ευχαριστώ το μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού που είπε πως ε, είναι σημαντικό η σωστή χρηματοδότηση. Θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη προσεχώς, το εάν θα διαθέσουμε δηλαδή επαρκή μέσα έτσι ώστε ο τομέα έρευνα και τη καινοτομία να έχει κεντρική σημασία. Έχει κεντρική σημασία για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον δεν αρκούν οι δεκάρικοι λόγοι, πρέπει να έχουμε γεγονότα. Κατόπιν, αναφέρεται και στην έκθεση το, θα πρέπει, το ότι θα πρέπει να δούμε αν χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τα μέσα μας. Πώς θα έχουμε απλοποιημένη διαδικασία, ταχύτητα, πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Πώς θα ξεφύγουμε από αυτό τον λαβύρινθο για να έχουμε μεγαλύτερες, ε, με περισσότερη απλοποίηση και ισχυρότερες δομές. Καμιά φορά, ξέρετε πως ούκεν το πολλό το εφ λιγότερα μέσα, περισσότερη ενίσχυση θα είναι το ε, καλύτερο αποτέλεσμα. Και βέβαια εδώ πέρα παίξει ένα σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και να μην ξεχνάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να βρούμε μια λύση για τις χώρες οι οποίες δεν θα έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο της αριστείας που απαιτείται για να χρηματοδοτηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας πραγματικός ανταγωνισμός για να δημιουργήσουμε ε, και σε μειονεκτικές περιοχές ε, κορυφαία ερευνητικά κέντρα. Αυτό ακόμα δεν έχει λυθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πυρίλο για ένα λεπτό. Χωρίς ε, μικρόφωνο ο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 θα πρέπει να αποτελέσει σημαντική, σημαντικό και όθηση, να δώσει μάλλον σημαντική όθηση στην εθνική ερευνητική προσπάθεια. Το εύρωμο πρόγραμμα για την έρευνα είναι πιο ευνοϊκό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν βελτιώθηκε το ποσοστό συμμετοχής του. Η δεν πέτυχε το στόχο. Όπως ε, σωστά λέγεται στην έκθεση της συναδέλφου Ματίας, χρειάζεται να υπάρξουν μέτρα διοικητικής απλοποίησης και μείωση των απαιτήσεων ε, Ελπίζω επίσης σε μια ευρεία συνεργασία και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά και εθνικά καθεστώτα χρηματοδότησης, ώστε να μην υπάρξει επικάλυψη και να υπάρξει βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τρέιτσακ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θέλω να σας πω ότι είναι φανερό πως ε, η καινοτομία αλλά και η τεχνολογική πρόοδος είναι οι ατμομηχανές για την ε, οικονομική επιτυχία και ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, εγώ όμως, όσον αφορά την έκθεση αυτή, μπορώ εδώ να διακρίνω δύο στοιχεία, δύο τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Πρώτον, Οι δυνατότητε τη αγορά, όπω επίση και οι κατάσταση επιχειρήσεων, θα μα οδηγούν στο ότι δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιου είδου ε, προποθέσει όσον αφορά την χορηγία κάποιων επιδόσεων. Ε, το κέρδο στην αγορά θα πρέπει να είναι το κριτήριο. Το κέρδο δεν είναι κάτι ε, για το οποίο δεν πρέπει να ντρέπεται κανεί. Το κέρδο είναι το μηχανή, το κέρδος είναι το κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη. Δεν έχω να σα πω τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Στερό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίω θεωρώ ότι είναι κάτι το θετικό το να προβαίνει κανεί σε επενδύσει για έρευνα και τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά όμω, δεν θα πρέπει να είναι και αυτή η πολιτική. θα πρέπει να εξετάζεται αλλιώς το ποιος θα ενισχυθεί. Δεν είναι τώρα μια κεντρική αρχή να καθορίζει προς τα πού θα κινηθεί ε, η έρευνα. Θα πρέπει όλοι να έχουν την ίδια δυνατότητα προσβάσεως εις την οικονομική ενίσχυση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι θα παίρνουν τα ίδια χρήματα. Επίσης άλλο καινοτομία και άλλο περιφερειακή πολιτική. Διότι δεν θα πρέπει τα προγράμματα και σχέδια τα οποία δεν αξιόλογα ε, να συγκρίνονται, να είναι στο ίδιο καλάθι με τα αξιόλογα. Άρα δεν θα πρέπει με τίποτα να λέμε ότι η κοινωνική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική, η γεωγραφική ανακατανομή της χρηματοδότησης ε, θα γίνεται με τα κριτήρια που προανέφερα, διότι αλλιώς θα έχουμε στρέβλωση στην αγορά της καινοτομίας. Η κυρία Σαρτόρη για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Ματίας για τη δουλειά της. Από την άλλη πλευρά μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί της και σε άλλα θέματα όπως αυτό της και τα ε, τα παραποιημένα έργα και πάντοτε η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω πως το γεγονό ότι η Κομισιόν τονίζει το θέμα τη καινοτομία και όχι μόνο τη έρευνα ε, είναι ένα σημαντικό μήνυμα, έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να ζητάμε τα σωστά πράγματα, αυτό που θύμισε και η Επίτροπο και που ε, σημαίνουν τελικά πιο σημαντικά κονδύλια, επί των οποίων ε, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αγωνιστεί. Ε, μια πεποίθηση ότι στο ε, πλάι της λέξης έρευνα θα πρέπει να υπάρχει πάντα και η λέξη καινοτομία. Ε, καινοτομία σημαίνει ακριβώς αυτόν τον τομέα που σημαίνει ε, ότι τα προϊόντα της έρευνας ανταποκρίνονται και στη ζήτηση της αγοράς. Και τρίτο θέμα το οποίο τονίζεται είναι η απέτηση που έχει η Ευρώπη να συνεχίσει να διατηρεί και να βελτιώνει το θέμα της ε, αριστείας και από την άλλη πλευρά να αφιερώνει ένα κομμάτι των πόρων της σε μια έρευνα πιο κοντινή στους πολίτες της επικράτειας, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, Εννοούμε πως πρόκειται για ένα επίπεδο από το οποίο μπορεί να προκύψει η εξαιρετική ιδέα, η ευφυής ιδέα που ανέκαθεν χαρακτήριζε τον κόσμο της έρευνας και των εφευρέσεων. Θα πρέπει λοιπόν όσοι πια έκαναν καλή δουλειά να μπορέσουν να βοηθηθούν όταν θα έχουμε τα κατάλληλα κονδύλια και το θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα κριτήρια της ε, ε, απλοποίησης διαδικασίας και στην ταχύτητα της επικύρωσης των προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Έντσου για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Το νέο στρατηγικό, κοινό στρατηγικό πλαίσιο που προτείνεται ε, από την απλοποίηση της διαδικασίας και την αύξηση της διαφάνειας μπορεί να διευκολύνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τα προγράμματα και τη χρηματοδότησή τους. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πτυχή που ίσως συζητάμε λιγότερο και να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονό ότι ο κ. Ρόλ, πρόεδρο τη Επιτροπή Ήτρε, το ανέφερε ήδη εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κρατών μελών γνωρίζει τεράστιε διαφορέ όσον αφορά τι ερευνητικέ και τι καινοτόμε δυνατότητε που έχουν οι διάφορε χώρε, τι ερευνητικέ υποδομέ και τι βιομηχανικέ υποδομέ. Γι' αυτό και θεωρώ πω το σημερινό πρόγραμμα χρηματοδότηση είναι ε, πλεονεκτικό για τι χώρε που είναι πιο προηγμένε. Και άρα οι διαφορέ δεν θα κάνουν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αυξηθούν. Γι' αυτό και πιστεύω πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να εντετικοποιηθεί η συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και η ε, χρηματοδότηση για την συνοχή να είναι ε, συμπληρωματική για το μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο. Και έτσι τα κράτη-μέλη που ε, είναι αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να ε, αναπτύξουν αποτελεσματικά και ενδιαφέροντα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Φόρντ, η κυρία Φόρντ, με για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Εισηγήτρια, συμφωνούμε πως η χρηματοδότηση της έρευνας μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως η υγεία, η γύρανση, η ενέργεια και η ασφάλεια τροφίμων. Και συχνά μένουν οι ανακαλύψεις στο εργαστήριο ή τις εκμεταλλεύονται άλλοι. Με την συνεργασία με την βιομηχανία έχουμε ενθαρρύνει μεγάλες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και ένα ισορροπημένο πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίξει και τις μικρές εταιρείες και με μεμονωμένες εστίες αριστείας αλλά βεβαίως θα αναγνωρίζει και το ρόλο μεγάλων εταιρεών και κορυφαίων πανεπιστημίων. Και βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να περιορίζονται εδώ πέρα τα προγράμματα της Ένωσης. Λιγότερα έντυπα, οπωσδήποτε περισσότερη απλοποίηση και περισσότερη έρευνα. Ε, η Επίτροπος συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με επιστήμονες στην περιοχή μου που είχαν αντιρρήσεις για την ε, αμεροληψία της, ε, του ελέγχου από συναδέλφους τους. Και βεβαίως δεν είμαι υπέρ του να βγάζουμε διάφορα νούμερα από το κεφάλι μας όσον αφορά τα στοιχεία αυτά. Σας ευχαριστώ. Γιόρταν σε για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να σας πω για τη χρηματοδότηση, διότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση να αυξηθεί. Επανειλημμένα, ακούστηκε σήμερα εδώ, ότι τα 80 δις αποτελούν σημαντική αύξηση της πληκοδότησης όμως δεν συμφωνώ 100% με αυτό διότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το 8ο πρόγραμμα με το αυτό το οποίο συζητούμε. Γιατί τώρα θέλουμε να καλύψουμε και ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Το Ίδρυμα για Τεχνολογία και, για τεχνολογία και Καινοτομία Έχουμε και επιπλέον γραμμή του προπολογισμού, οπότε εάν μετά τις διαπραγματεύσεις οι πόροι για την έρευνα συρρυκνωθούν, τότε διατηρώ σημαντικές επιφυλάξεις όσον αφορά τις προτεραιότητες που θέλουμε να τάξουμε. Όσον αφορά τώρα πάλι την ε, γεωγραφική κατανομή. Συχνά λέμε ότι τα βασικά κριτήρια για την επιλογή είναι η επιστημονική αριστεία. Όμως θα πρέπει αυτή να οριστεί με τρόπο που να μπορεί να ε, είναι εφαρμοστέα στην πράξη. Δεν θα πρέπει αυτό να είναι αποκλειστικότητα των, ε, των πολύ πιο μεγάλων ε, σχεδίων και προγραμμάτων των πολλών εκατομμύριων. Θα πρέπει το πρόγραμμα πλαίσιο να καλύπτει όλα τα μεγέθη προγραμμάτων και έργων να εξετάζεται επομένω ε, η ποιότητα ε, για τις περιφέρειες και για τα κράτη-μέλη και βέβαια μιλούμε τώρα για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Κατακλείθηκε το σχετικό συμβούλιο συμφωνεί ότι συνήθως ε, τα πιο γνωστά πανεπιστήμια και πιο μεγάλε χώρε ωφελούνται από αυτό το πλαίσιο. Άρα, να μην το λέμε ideas, ιδέες, να το λέμε fame, fame, fame όπως το serial. Το έργο, εν πάση τόσο, θα πρέπει ακριβώ να είναι και ω κριτήριο το κατά πόσο ένα σχέδιο ε, επιδέχεται την υλοποίηση του εύκολα. Τι κάνω, ένα λεπτό. Ε, αντιμετωπίζουμε κρίση και η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, η παιδεία ε, η τεχνολογία είναι μέσα πολύ σημαντικά για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και πρόθεση τη οικονομία. και γι' αυτό και οι διαδικασίε πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα για χρηματοδότηση θα πρέπει να απλοποιηθούν. Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την καινοτομία και την τεχνολογία θα πρέπει να βασιστεί σε συντονισμό των προγραμμάτων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη και να επιτρέψει να βρεθούν λύσει για τι δημογραφικέ αλλαγέ για το γεγονό ότι πρέπει να διαχειριστούμε με βιώσιμη βιώσιμο και ισότιμο τρόπο του πόρους μα και επίση θα πρέπει να στηριχθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ. Και αυτή η συμμετοχή θα πρέπει να είναι πάνω από το 15%. Γι' αυτό και η απλοποίηση και η άρση των γραφειοκρατικών φραγμών είναι ουσιώδη ώστε να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε τι οικονομικέ δραστηριότητε. Χρειάζονται επιπλέον δε πόροι για τι εφαρμογέ όπω το πρόγραμμα Γαλιλαίο που πρέπει να να λειτουργήσει στο maximum. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαρσινκέβιτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ησυχήτρια για τον συμβασμό τον οποίο επέτυχε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούμε με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας ε, κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ένα στρατηγικό πλαίσιο το οποίο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ε, στον κόσμο. Επίσης καλωσορίζουμε την ιδέα της απλοποίησης των ε, διαδικασιών Υπάρχουν διαφορές πράγματι μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο της έρευνα και τη καινοτομία και της πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα. Υπάρχει ένα χάσμα, εάν θέλετε, μεταξύ των λεγόμενων παλαιών και καινούριων κρατών μελών απλοποίηση και η εναρμόνιση των διαδικασιών είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ε, διαφανούς ευρωπαϊκής ερευνητικής ζώνης και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το χαμηλό επίπεδο εκπροσώπησης κάποιων περιφερειών το οποίο θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με την ε, βελτίωση πραγμάτων όπως η δυνατότητα ενσωμάτωσης. Καλωσορίζω επίσης ε, την διασυνοριακή έρευνα, αλλά νομίζω πως η συζήτηση βεβαίως αφορά κυρίως τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κορέιο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρία Ματία για την εξαιρετική τη έκθεση σημασία του κοινού στρατηγικού πλαισίου για την χρηματοδότηση τη έρευνα και τη τεχνολογία. Ξεπερνά του αυστηρά επιστημονικού στόχου. Είναι ένα ζωτικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020, για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία απασχόληση, για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Αλλά πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν και τα, και τα σφάλματά θα πρέπει να ε, υλοποιηθεί αυτό το πράγμα μεγαλύτερη φιλοδοξία και ακρίβεια για να μπορέσουμε ταυτόχρονα να ε, εξαπλώσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ε, στην κοινωνία και στην οικονομία. Να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε ακούραστα να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε στις προσπάθειες συνεργασίας, να προωθήσουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας όπως ήδη τονίστηκε μέχρι τώρα δύο διαφορές, δηλαδή να μειωθούν ε, οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πολλή δουλειά πρέπει ακόμα να γίνει, πρέπει να ε, παγιωθούν οι δρόμοι της αριστείας. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε σε αυτό μας το στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω πως η κυρία Τόγια δεν είναι στην αίθουσα. Και άρα ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Υπάρχουν 12 που ζήτησαν το λόγο. Εάν τηρήσετε το χρόνο θα δώσω το λόγο σε όλους. Ξεκινάμε με τον, την κυρία Αντωνέσκου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ την ε, κυρία Ματίας για την εξαιρετική της έκθεση. Ε, ε, κυρίως ε, για εκείνα τα κράτη-μέλη που είναι πιο πίσω στην καινοτομία που υστερούν γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διαφορές στην χρηματοδότηση που αντικατοπτρίζονται στη συμμετοχή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και πιστεύω πως χρειαζόμαστε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, έναν μηχανισμό που να μπορέσει να εξισορροπήσει αυτή την κατάσταση και να ενισχύσει τις δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα κρατημέλη. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν ήταν ε, αρκετές. Ακόμα και αν υπάρχουν σημαντικά μέσα για την ε, αναζωγόνηση των οικονομιών μας, ε, χρειαζόμαστε νέες προσεγγίσεις και αυτό θα πρέπει να, είναι, να γίνει μέσα στη νέα προγραμματική μας περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστηκαν διάφορα ενδιαφέροντα ζητήματα και χάρηκα για αυτό το οποίο είπε η κυρία Επίτροπος για σημεία που πρέπει να τονίσουμε στο μέλλον. Δεδομένης κατάσταση ε, στην Ευρώπη Ξέρετε πως μας είπαν διάφοροι οικονομολόγοι πως ε, καλό είναι να συμμαζευτούμε αλλιώς θα καταρρεύσουμε. Οπότε μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε δουλειές και ανάπτυξη και έρευνα και καινοτομία θα παίξουν εδώ πέρα σημαντικό ρόλο. Οπότε θεωρώ πως έχει δίκιο η Επίτροπος όταν λέει πως πρέπει να δώσουμε βάρος στην ε, απλοποίηση, μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στις γυναίκες και να είμαστε πιο κοντά στι προκλήσει τη κοινωνία και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα γιατί δεν έχει νόημα να κάνουμε έρευνα για τόσο ωραία θέματα όπως παραδείγματος χάρη σεξουαλική ζωή των βατράχων εάν δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα σε θέσεις εργασίας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Μπασέσκου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έρευνα, η παιδεία, η καινοτομία είναι τα βασικά στοιχεία μιας ανταγωνιστικής και ισχυρής οικονομίας. Σε ένα δύσκολο πλαίσιο είναι ε, επίσης σημαντικά για να μπορέσει να ε, κινηθεί και πάλι μια βιώσιμη οικονομική. Γι' αυτό και χαιρετίζω το πράσινο βιβλίο της Κομισιόν που είναι ακόμα πιο σημαντικό μέσα σε αυτή την περίοδο. Και βλέπω ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην μείωση των διαφορών ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τη χώρα μου. Αυτή η πτυχή είναι πολύ σημαντική. Γιατί, ε, δεν γιατί έχουμε ποσοστά πολύ χαμηλότερα από όλα τα άλλα κράτη, τα ευρωπαϊκά, για σχεδόν όλους τους δείκτες. Στην κατάταξη για την καινοτομία η Ρωμανία είναι κάτω από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών. Ε, ταυτόχρονα θα ήθελα να τονίσω την περιφερειακή συνεργασία που ευνοεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ως προς αυτό η Ρωμανία έκανε μια πρόταση, δηλαδή τη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου προηγμένων μελετών για το σύστημα Δούναβης ε, ε, δέλτα του Δουνάβεως με την Μαύρη Θάλασσα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια και να παρακαλέσω την Επίτροπο ειδικά στα ζητήματα προϋπολογισμού να γίνει λίγο πιο φιλόδοξη είδαμε αυτή την αύξηση στα 80 δισεκατομμύρια, αλλά αυτό έγινε με τη συμπερίληψη πολλών άλλων προγραμμάτων, οπότε η καθαρή αύξηση ήταν μικρή. Οπότε με τα ίδια τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. τους πόρους του διοξιδίου του άνθρακα, δεν θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε προβληματικούς τομείς ε, ε, τους οποίους θα ορίσουμε από κοινού με τους Υπουργούς Οικονομικών για να πούμε πως αυτά τα λεφτά πάνε μόνο σε προγράμματα α, κοινής ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας, οτιδήποτε εισπράξουμε από τον φόρο του άνθρακα. Θα προσπαθήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο, κυρία Πρόεδρε, μαζί με το δημοσιονομικό πλαίσιο βεβαίως. Νομίζω πως θα μπορούσε να μας βοηθήσει βραχυπρόθεσμα για την έρευνα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ζήτημα αυτό για να αναπτύξουν ανάλογες υπηρεσίες για να έχουμε και μια μελλοντική στρατηγική για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλτασάρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ αργά προχωρά στον τομέα της επιστήμης. Δεν μπορεί να κερδίσει την ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία. Τα 27 μέλη, κατά μέσο όρο επενδύουν μόνο το 2% του ΑΕΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη αντί να σεβαστούν τον στόχο του 3% που έχει θέσει η Κομισιόν. Φέρεται λοιπόν σκόπεμη η δημοσίευση του πράσινου βιβλίου από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα επιτρέπει να ξεκινήσουμε ενεργά τη συζήτηση όπω προκύπτει και από την εξαίρετη έκθεση που εκπώνησε η συνάδελφος Ματίας. Σημερίζομαι το αίτημα της εισηγήτριας σε σχέση με τη δημιουργία ενός κοινού πανευρωπαϊκού ταμείου που στόχο θα έχει την προώθηση της ε, συνεργασίας στην έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μειωθούν οι ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό κάθε μέτρο να, να... κάθε μέτρο να προηγείται ένα μια ανανέωση του πλαισίου για το 2014-2020. Σας ευχαριστώ, κύριος Ματούλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έρευνα και καινοτομίας είναι η συνθήκη των ΟΝΟΥ ΚΑΝΕΦ να προχωρήσουμε όμω πρώτα από τα χρειάζονται περισσότεροι πόροι προεκοδότηση ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε το 3% του ΕΕ, το οποίο θέλουμε να καταλαμβάνει η έρευνα και η καινοτομία. Μέχρι το 2020 όμω ακόμα υπάρχουν φραγμοί σε αυτό το στόχο για την υλοποίησή του, διότι βασικά όσον αφορά ε, τις εθνικές αρχές αλλά και τις περιφερειακές αρχές υπάρχουν ε, στατικές τώρα που ε, ε, χρειάζονται από, από κατάτμιση, από επικαλύψεις Επομένω χρειάζεται μια κοινή στρατηγική για έρευνα και καινοτομία τόσο ώστε να, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε ομοθετικά τη χρηματοδότηση και αυτό θα να γίνει με κάποιες ε, πιο απλές δομές πιο αποτελεσματικού μηχανισμούς και έτσι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα βασικά όργανα χρηματοδότησης και ή στην συνέχεια να μπορούμε να προχωρήσουμε σε επίπεδο κρατών μελών, τοπικών αρχών και να προχωρήσουμε με τρόπο συνεπή. Και άρα η χρηματοδότηση να ε, καλύψει την ιδιωτική επένδυση <clears throat> και να μπορέσουμε να τονώσουμε πάλι την συμμετοχή των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτά τα έργα και προγράμματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία, ο κύριος Γκουτιέρες. Α, συγγνώμη. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ και την κυρία Ματία για την εκθεσή τη και εγώ θέλω να πω στην κυρία Επιτρόπο τα εξή. Πρώτα πρώτα μην ξεχνάτε τα μικροπρογράμματα, διότι από εκεί ξεκινάμε. Είναι η βάση. Τα χρειαζόμαστε ούτω ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα μικρά πανεπιστήμια. Δεύτερον, νομίζω ότι αυτό το οποίο λείπει εδώ είναι ανθρώπινη πόρη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα υποτροφιών, ούτω ώστε τα μεγάλα πανεπιστήμια, τα μεγάλα ιδρύματα να έχουν όλα ένα και περισσότερου ε, υποτρόφου. Άρα θα πρέπει να δώσουμε λιγότερη σημασία στα κτίρια. Χρειάζονται λιγότερες, λιγότερα κτίρια. Χρειάζεται να τονώσουμε τους ανθρωπίνους πόρους. Άρα θα σας βοηθήσουμε. Αλλά όμως θα πρέπει <clears throat> να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες απλουστευτικές, απλούστερες. Θα πρέπει επομένω να έχουμε κάποια διαφάνεια στις διαδικασίες από πλευράς ε, των κρατών μελών και θα πρέπει να δεσμευτείτε προς τούτο και έτσι εμείς θα σας ε, υποστηρίξουμε απερίφραστα 100% αλλά θα πρέπει να προχωρήσετε προς μια τέτοια πρόταση απλούστευσης να την βάλετε ή στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ λέει πρώτος και τώρα. Ο κ. Ματίας. Η κυρία. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια. συζητάμε και συζητάμε για την ε, ανάπτυξη και ε, θα έπρεπε να μιλάμε για την ανάπτυξη περισσότερο από όσο μιλάμε για την κρίση. Δεν γίνεται όμως κάτι τέτοιο, διότι τα της ανάπτυξης και τα της καινοτομίας δεν αποτελούν φαίνεται προτεραιότητα, υψίστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως εσείς κύριε Επίτροπε διαφωνείτε, αλλά μόνο εσείς διαφωνείτε. Και άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει προς χάρη όλες τις ε, κοινωνίες χρειάζεται να τονώσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα. Θα πρέπει να πάει παντού η ανάπτυξη. Θέλουμε απλούστευση. Θέλουμε λιγότερη γραφειοκρατία, ευκολότερη προσβασιμότητα στην χρηματοδότηση και θέλουμε μη ε, χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά δεν αφορούν οι επιχειρήσει αυτέ το δικό σας ε, χαρτοφυλάκιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ε, ευμενή ιστορική αγορά και να υπάρχει κατάλληλο πλαίσιο ώστε να μπορούν οι εμπλεκόμενοι όλοι να συνεργαστούν. Δεν Η κυρία Νταντσίλα, ξέρουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχους να αυξήσει τις δαπάνες για την καινοτομία και την έρευνα μέχρι το 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι το 2020. Όμως όλα τα κράτη-μέλη δεν θα τα καταφέρουν να πετύχουν αυτό το στόχο. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση ολοκληρωμένη και αυτό μέσα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, ούτως ώστε οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις να γίνουν στην πράξη ως μέλος ε, της Επιτροπής ε, Γεωργίας θεωρώ πως το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν, θα πρέπει να συνδυάσει ε, τις διάφορες συνεργασίες μέσα στο, κοινό, στο πλαίσιο κοινής ε, πολιτικής ε, και ταμεία συνοχής, ε, διαρθρωτικά ταμεία, ώστε να μπορούμε να βασιστούμε σε όλα τα προγράμματα που υπάρχουν και να ενθαρρύνουμε έτσι την έρευνα και την ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Να αναπτύξουμε τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες καινοτομία των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Όταν μιλάμε για την έρευνα και ενοτομία θα πρέπει να θυμόμαστε πως στόχος είναι η πρόθεση ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η δημιουργία θέσεων εργασίας. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε καλύτερη έρευνα. Οι επιχειρήσεις ε, πρέπει να αποτελέσουν τμήμα της ερευνητικής κοινότητας και να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε σε κορυφαία έρευνα αλλά και να επενδύουμε σε πρακτική καινοτομία. Και όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να στηρίξουμε και βεβαίως έχουμε και τα διαρθρωτικά ταμεία για το σκοπό αυτό. Οπότε μπορεί να μειωθεί το κατόφλι για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα πλαίσιο. Σας ευχαριστώ, Όμπερ Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εάν δούμε το πόσο έχουμε προχωρήσει όσον αφορά την έρευνα και το ποια είναι η προσθέμενη αξία παράγεται, διαπιστώνουμε το εξή. Στην ε, Ευρώπη έχουμε μετατοπίσει την παραγωγή σε άλλες χώρες και εδώ πέρα υπάρχει μόνο το marketing. Οπότε μειώνουμε συνεχώς τις βιομηχανικές μας δυνατότητες και οδηγούμαστε όλο και βαθύτερα στην ύφεση μεγάλα έργα όπως ε, ο Γαλιλαίος εντωμεταξύ θα πρέπει να έχουν δική τους γραμμή του προϋπολογισμού και να μην προσθεθούν στο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός σχετικός ε, και με διαρθρωτικά ταμεία και να χρηματοδοτήσουμε όλες τις σχετικές επενδύσεις αλλά αρκεί να κάνουν και τα κράτη-μέλη βεβαίως αυτό που τους αναλογεί και να μην ξεχνούν και τα κριτήρια τα ποιοτικά σας. Ευχαριστώ. Μπρόντς. Είναι αυταπόδεικτο ότι η έρευνα και η ανάπτυξη θα πρέπει να διευκολυνθούν σε όλα τα κράτη. Όλα ένα περισσότερο είναι αναγκαία από τη στιγμή που η οικονομία μας υπόκειται αθέμητο ανταγωνισμό από τις ε, χαμηλόμιστες οικονομίε. οικονομίες. Ο μόνος τρόπος ο αναπτυσσόμενος κόσμος να ανταγωνιστεί με τις, ε, τους, είναι να μπορέσει να, ηγηθεί στις νέες τεχνολογίες οι καρποί αυτή τη έρευνα θα πρέπει να προστατεύονται από ένα αποτελεσματικό σύστημα ευρεσιτεχνιών. Δεν θα πρέπει να μπορούν ε, ατιμωρητοί να ε, αντιγράφουν τις εφευρέσεις του δυτικού κόσμου να αναδυόμενες χώρες. Πρόσφατα ε, παραγωγή της από Ανατολής ήταν στα δικαστήρια λόγω της ε, αντιγραφής διαφόρων ε, προϊόντων που είχαν κατασκευαστεί στο Μόναχο. Σας ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση, η κυρία Μπέρκμαν. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαίρω και εγώ την κυρία Ματίας για την έκθεσή του. Ε, η Ευρώπη είναι η πλωσεότερη περιοχή στον κόσμο, αλλά είπα ε, η Ιαπωνία και άλλες χώρες επενδύουν πολύ περισσότερο σε έρευνα και ανάπτυξη. Οι επενδύσεις στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, αλλά όσον αφορά το στόχο του 2020 για ένα συνολικό ποσό 3% του ΑΕΠ, μόνο 6 χώρες το έχουν φτάσει. Έχουν περάσει αυτή τη στιγμή το 2% της 100, οπότε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις κοινωνικές Πτυχέ ε, της υπόθεση αυτής. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ειδικά την πτυχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των γυναικών επιστημόνων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η Επίτροπος Ιέγαν Κουίν. Η Επίτροπος. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ με ενθαρρύνει η συζήτηση, τα όσα ακούστηκαν εδώ. Άκουσα και τον κύριο Ρούμπιχ και, οι άλλοι σα γίνεται τον προπολογισμό. Βεβαίω, ε, επειδή με επαφή σε εσά αλλά και στο Συμβούλιο και κατόπιν των όσων ακούω σήμερα θα είναι σύμμαχο σημαντικό μου για την αύξηση τη πληροδότηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, <clears throat> κατακλείδη να δούμε πώ θα οργανώσουμε την πολιτική μα συνόψη του 2020. Θα πρέπει να περιστρεφόμαστε δύο από τρει ε, αλληλοσχετιζόμενου άξονε σε σχέση με προτεραιότητε. Πρώτον, αριστεία στα επιστημονικά και δεύτερον να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές προκλήσεις σε σχέση με αυτό που έχουν επισημανθεί την πολιτική του και τρίτος άξονας ηγεμονία, πρωτοπορία, βιομηχανική βοήθεια σε επιχειρήσεις και βοήθεια στην καινοτομία. Ξέρω ότι κυρία Ματίας αυτοί οι άξονε δεν αντιστοιχούν στα τρία σα κεφάλαια. Νομίζω όμω ότι έχουμε την ίδια βάση για του ίδιου στόχου. Να έχουμε απλώ τη διαδικασία, να έχουμε πρωτοτυποποίηση τη. Ε, και να έχουμε επίσης και συγκεκριμένο προγραμματισμό για την, για την ε, χρηματοδότηση και να έχουμε ε, κανόνες κοινούς και επίσης να έχουμε περισσότερη εξωτερήκευση να έχουμε μείωση των δαπανών και να έχουμε μια προσέγγιση της επιστροφής των εξόδων. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τον φορμό ομοιογένεια στην λογιστική των ε, συμμετεχόντων και επίσης να δούμε πώς θα γίνει με τις ε, φάπαξ προζημιώσεις. Χρειάζονται και επίσης ε, κάποιες οδηγίες με τις μονοπευθυντικές θηρίδες, με websites και λοιπά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε τους στόχους μας για τον ορισμό του 2020 να έχουμε συνέργεια, να έχουμε συμπληρωματικότητα. Το ορίζοντα του 2020, το, πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να βοηθήσει παντού, ε, να πρέπει τα ταμεία συνοχής να βοηθήσουν ε, τη δημιουργία δυνατοτήτων μας, δυνατοτήτων μας και τις επιλέξιμες περιοχές. Το Περιφερειακό Ταμείο θα πρέπει να βοηθήσει τις στρατηγικές, τις εξειδίκευσεις επί τη βάση του στόχου της ε, βοήθειας της αριστείας και επομένω, θα κατεβάσουμε προτάσεις με το τέλος ενεστώτος έτου, Οι προτάσεις μας ε, που βοηθήθηκαν πάρα πολύ από την έκθεσή σα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα όσα είπατε στην έκθεση και άρα εμεί θα τα μελετήσουμε περαιτέρω, σοβαρά και εγώ η Ιδία αλλά και οι συνεργάτε μου ε, τι επόμενε μέρες. Σα ευχαριστώ Επίτροπε. Τώρα το λόγο έχει η εισηγήτρια, η κυρία Ματίας, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία, Επίτροπε, ε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλα τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ε, επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χρέλ να πω ότι Ήδη αυτή η έκθεση είναι το κομμάτι ενός συνόλου εκθέσεων και όπως η έκθεση Καρβάλιου, Μέρκελ, Οντί, ε, αλλά είναι ένα σύνολο που, ε, εκθέσεων που προχωρούν προς την ίδια κατεύθυνση και πιστεύω πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά από τη συζήτηση που έγινε. Υπάρχει όμως και ένα σύνολο προσανατολισμών του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θα ήθελα η Κομισιόν να λάβει υπόψη όλα αυτά τις συστάσεις του οίκου της Δημοκρατίας Μιλάμε για το τρίτο μεγαλύτερο στρώμα χρηματοδότησης ε, μετά από την ε, γεωργία ε, και είναι πολύ σημαντικό για να αναπτυχθεί η ποιοτική απασχόληση, να ξεφύγουμε από αυτή την πληγή που είναι η επισφάλεια των ερευνητών, κυρίως των νέων ερευνητών, είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε. Και μια άλλη διάσταση που θα ήθελα να δούμε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν μπόρεσα να αναφερθώ σε όλες ε, και γι' αυτό και εστιάζεται την προσοχή μου σε αυτά. Είχαμε και μια Ευρωπα... Είχα και μια πρόταση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης. Έχουμε μια συμβεβαιστική λύση ώστε να έχουμε ένα ειδικό κλάδο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως που ήδη υπάρχει και ελπίζουμε ότι η εθνική χρηματοδότηση, ε, η δημόσια χρηματοδότηση, να σκεφτόμαστε σε τι χρησιμεύουν για τις ερευνητικές μονάδες, για τα πανεπιστήμια, για άλλους εταίρους, για να εξυπηρετήσει επιχειρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε σε αυτό το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο την ενίσχυση της, ε, των επενδύσεων σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30. Τώρα, σύμφωνα με την μερίσια διάταξη, πρέπει να συζητήσουμε την ε, σύσταση της κυρίας Κοπά για την ανταλλαγή των ε, ε, γεωρικών και ελευτικών προϊόντων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παλαιστίνη.